Συνεχίζουμε τις ψηφοφορίες. Έκθεση Ριβαζή. Έχει το λόγο η συγκίτρια αν το επιθυμεί. Ευχαριστώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, η έκθεση αυτή αφορά τον έλεγχο των ραδιενεργών ουσιών που περιέχονται στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης, το πόσιμο είδωρ για να εξασφαλίσουμε μια συνοχή του κειμένου και μετά από διαβουλεύσεις με τις υπηρεσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τις πολιτικές ομάδες ήθελα να κάνω μια τεχνική τροποποίηση στη δεύτερη τροπολογία για να διαγραφεί το εξή. Μετά από την παραπομπή του νομοθετικού ψηφίσματος στη, στα Εθνικά Κοινοβούλια και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών. Και μετά τη ψηφοφορία θα ήθελα να μου δώσετε για λίγο το λόγο προκειμένου να ε, στείλω ένα μήνυμα εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μάλιστα, 56 τροπολογίες έχουμε μαζί. Ψηφίζουμε ψηφίσουμε ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνονται. Ψηφίζουμε την πρόταση της Επιτροπής. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, Παρακαλώ, σηκώνετε τα χέρια σας γιατί δεν καταλαβαίνω. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίνεται. Και με ονομαστική κλίση, ψηφοφορία για το σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος, άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται και το νομοθετικό ψήφισμα και παρακαλώ την εισηγήτρια να λάβει το λόγο. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε και ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη σας. Είναι πραγματικά σημαντική αυτή η ψηφοφορία. Εκ μέρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα ήθελα να απευθύνω έκκληση προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διαβιβάσει τροποποιηθήσα έκθεση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στα Εθνικά Κοινοβούλια και στην Επιτροπή των Περιφερειών για να ξαναρχίσει η νομοθετική διαδικασία με βάση τη διαδικασία τη συναπόφαση. Η πρόταση της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι μια ε, δημοκρατική ανοησία. Δεν έχει κανένα νόημα και φάνηκε και στην ψηφοφορία μας στην αρμόδια επιτροπή. Ευχαριστώ θερμά τους συναδέλφους. Η έκθεση αφορά τον έλεγχο των ραδιενεργών ουσιών που εμφανίζονται στο πόσιμο είδωρ. Πρόκειται για ένα ζήτημα δημόσια υγεία. Θα πρέπει λοιπόν και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να αναμειχθεί στην νομοθετική διαδικασία. Γιατί με τη δράση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή στερεί από του Ευρωπαίου πολίτε τη δυνατότητα συμμετοχή σε μια δημοκρατική συζήτηση και ψηφοφορία. Δεν είναι θέμα αν είμαστε υπέρ ή κατά τη πυρηνική ενέργεια. Θέλουμε να προστατεύσουμε την ποιότητα του πόσιμου ύδατο, του ύδατο που καταναλώνουμε καθημερινά. Και η Ευρατόμ δεν είναι σε καμία περίπτωση η νομική βάση, η δόκη. Ω Ως εκ τούτου, και ολοκληρώνω, ε, επιβάλλεται η διαδικασία της συναπόφασης με βάση το άρθρο 192 της Συνθήκης της Λισαβόνας. Αυτή είναι η σωστή νομική βάση. Μάλιστα, πριν την έκθεση Κοζές, ζήτησε το λόγο ο Επίτροπος Ρεν. Παρακαλώ. κυρία Πρόεδρε, έντυπα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είναι μεγάλη σημασία αυτή τη στιγμή και αυτή τη ψηφοφορία για το οικονομικό μέλλον τη Ευρώπη. Είναι κάτι το οποίο δεν μπορώ να το τονίσω αρκετά. Μαζί με το εξάπτυχο, οι δύο αυτοί οι κανονισμοί μας φέρνουν σημαντικά βήματα προς μια οικονομική και νομισματική ένωση Θέλω να χρησιμοποιήσω την ευκαιρία για να ευχαριστήσω όλους τους εισηγητές, σκιώδεις εισηγητές, άλλους βουλευτές, φίλους και συναδέρφους που έχουν συνεργαστεί μαζί με την Κομισιόν και την Προεδρία του Συμβουλίου για να μπορέσουμε να κάνουμε πραγματικότητα αυτό το νομοθέτημα. Θέλω να σας ευχαριστήσω επίσης όλους για τις πολλές τροπολογίες που έχετε εισαγάγει. Πολλές φορές με την επιμονή που δείχνει ακόμα και ξεροκεφαλιά και που τελικά όμως έχουν ενισχύσει τις προτάσεις στη διαδικασία αυτή την νομοθετική. Τολμώ να πω ότι αν το εξάπτυχο και το δίπτυχο, το six-pack και το, δι... το two-pack ήταν πραγματικότητα στην αρχή της δημιουργίας του ευρώ, δεν θα είχαμε ποτέ να αντιμετωπίσουμε μια τέτοια κρίση ή τουλάχιστον θα είχαμε ξεπεράσει την κρίση πολύ πιο γρήγορα και με λιγότερο οικονομικό και κοινωνικό κόστος. Με τη σημαίνει ψηφοφορία θα καταδείξουμε πιστεύω σε όλους τα ωφέλη και τη λειτουργία της κοινωτικής μεθόδου. Αν δούμε με τη χρονική απόσταση το πώς εξελίχθηκε η κρίση και επίσης αν δούμε την επιμονή της Κομισιόν για ένα ταμείο εξάλληψης του χρέους, εγώ μόναχα να ελπίζω μπορώ ότι το Συμβούλιο θα είχε υποστηρίξει την κοινοτική μέθοδο και τις προτάσεις της Κομισιόν ήδη από την άνοιξη του 2010, πριν από τρία χρόνια. Αναφέρομαι στην Σύνοδο του ΕΚΟΦΗΝ 9 και 10 Μαΐου 2010, όταν η Κομισιόν την ημέρα της Ευρώπης σε μία από τις συνεδριάσεις μας για την αντιμετώπιση της κρίσης έκανε την πρόταση να δημιουργηθεί ένας ενιαίος μηχανισμός χρηματοπιστωτικής σταθερότητας στην Ευρώπη που να βασίζεται σε εγγύησεις του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ύψος 60 δισεκατομμυρίων και επίσης με κοινέ εγγύησεις των κρατών μελών πέραν αυτού. Με τον τρόπο αυτό θα είχαμε να θέχαμε το μεγάλο μπαζούκα όπως λέγεται το οποίο θα είχε δαμάσει τη χρηματοπιστωτική κρίση προτού να αναγκαστεί η ηγετική τράπεζα να προβεί στις μεγάλες χρηματοδοτήσεις προς την τράπεζα και το πρόγραμμα ε, οριστικών αγορών αξιογράφων. Τελικά μόνο πέρσι μπόρεσε αυτός ο θεσμός το ESM να δημιουργηθεί που έχει πλέον ισχυρό κεφάλαιο και μεγάλη δυνατότητα παρέμβασης. Νομίζω ότι θα είχαμε αντιμετωπίσει καλύτερα την κρίση και θα είχαμε δώσει ταχύτερα αποτελέσματα για τους πολίτες μας αν η αρχική πρόταση της Κομισιόν είχε γίνει πραγματικότητα τον Μάιο του 2010. Κύριε Πρόεδρε, νομίζετε ότι μπορώ να συνεχίσω. Σας ευχαριστώ. Το εκτιμώ ιδιαίτερα. Θα ήθελα να κάνω σαφές ότι οι προτάσεις της Κομισιόν σε σχέση με τα μελλοντικά βήματα ακολουθούν την εξής πορεία. Και θέλω και την υπομονή σας. Και συγχωρήστε με αν έχω μακρηγορήσει με τα δικά μου μέτρα αλλά πρόκειται για μια δύσκολη, εύθραυστη αλλά και πλήρη λύση για τα προβλήματα αυτά. Μετά από την έγκριση λοιπόν της νομοθεσίας που προτάθηκε η Κομισιόν για το δίπτυχο, η Κομισιόν προτίθεται να κάνει βήματα στο άμεσο μέλλον προς μια βαθιά και γνήσια ε, οικονομική και νομισματική ένωση. Μέσα σε 6 και 12 μήνες θα κάνουμε τα πρώτα βήματα για να υπάρξει το σχέδιο η ηλιοτυπία της Κομισιόν για μια ενιαία αντιμετώπιση με ένα ταμείο εξάλληψης του χρέους που θα είναι ένα σημαντικό στοιχείο για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στην πλήρη ένωση κάτω από συνθήκες αυστηρού ελέγχου. Το επόμενο βήμα θα είναι η αποκοινού θέση του κινδύνου που θα πρέπει να συμβιβάσει να συνοδεύει από πραγματική πειθαρχία στα επίπεδα του προϋπολογισμού και επίσης μια καλύτερη ολοκλήρωση των εργαλείων για τη χρηματοπιστωτική πολιτική θα πρέπει να συνοδεύεται από αντίστοιχες κινήσεις πολιτικής ενσωμάτωσης που να οδηγούν και σε μεγαλύτερη πολιτική λογοδοσία. Η Κομισιόν θα δημιουργήσει μια ομάδα εμπειρογνώμων, για να μπορέσει να εξετάσει τα θετικά και αρνητικά στοιχεία, τα εμπόδια, τις σωστές επιλογές για να μπορέσει να αντικατασταθεί η εθνική έκδοση χρέους από μια κοινή έκδοση χρέους με τη μορφή ενός ταμείου εξαλείψεως του χρέους και ευρώ ομολόγων. Η ομάδα αυτή θα έχει σαν εντολή να εξετάσει τις απαραίτητες νομικές πρόνοιες που θα πρέπει να ληφθούν, τη μορφή που θα πρέπει να έχει η χρηματοπιστωτική αρχιτεκτονική και το συμπληρωματικό πλαίσιο που πρέπει να συνοδεύει όλα αυτά. Το θέμα της, νομική, της ε, πολιτικής λογοδοσίας θα πρέπει να είναι ένα από τα βασικά στοιχεία αυτού του συστήματος. Η ομάδα αυτή σοφών θα λάβει υπόψη τη συνεχιζόμενη μεταρρύθμιση της ευρωπαϊκής δημοσιονομικής και οικονομικής διακυβέρνησης και θα εξετάσει και την προσθέμενη στη αξία για αυτά τα εργαλεία. Και η ομάδα επίσης θα δώσει ιδιαίτερη σημασία στις συνεχιζόμενες μεταρρυθμίσεις όπως είναι η εφαρμογή του μηχανισμού σταθερότητας, του διπτύχου και άλλων εργαλείων. Στην ανάλυση αυτή η ομάδα θα λάβει υπόψη τα θέματα βιωσιμότητας των δημοσίων οικονομικών της αντιμετώπισης του ηθικού κινδύνου και άλλα κομβικά θέματα όπως η χρηματοπιστωτική σταθερότητα και ολοκλήρωση, καθώς και η μετάδοση της νομισματικής πολιτικής. Τα μέλη της ομάδος θα είναι εμπειρογνώμονες στα οικονομικά, δημοσιονομικά θέματα, τα νομικά θέματα, τις χρηματοπιστωτικές αγορές και τη διαχείριση δημοσίου χρέους. Και η ομάδα αυτή θα παρουσιάσει την τελική της έκθεση προς την Κομισιόν πριν από το Μάρτιο του 2014. Η Κομισιόν θα αξιολογήσει το περιεχόμενο αυτής της έκθεσης και εάν αυτό είναι απαραίτητο θα υποβάλει προτάσεις πριν από το τέλος της εντολής της. Η διερεύνηση περαιτέρω τρόπων για να υπάρξει πρόληψη των χρηματοπιστωτικών κρίσεων και επίσης η δυνατότητα προγραμμάτων δημοσίων επενδύσεων ε, χαρακτήρα εφάπαξ με τη χρηματοδοτική συμφορά των κρατών μελών θα είναι κάτι το οποίο θα αντιμετωπιστεί το, την άνοιξη και το καλοκαίρι του 2013 στα πλαίσια του χρονοδιαγράμματος που δημοσίευσε η Κομισιόν για την σύγκληση σε οικονομικό επίπεδο. Μετά από την απόφαση που θα ληφθεί για το επόμενο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο για την Ευρωπαϊκή Ένωση και πριν από το τέλος του 2013 η Κομισιόν θα καταθέσει τις εξή προτάσεις για να βελτιώσει το πλαίσιο χρηματοοικονομικής διακυβέρνησης. Μέτρα για μεγαλύτερη εξάντε σύγκληση και συντονισμό των μεγάλων πολιτικών μεταρρυθμίσεων και οικονομικών μεταρρυθμίσεων και τη δημιουργία ενός εργαλείου σύγκλησης το οποίο θα δίνει και την χρηματοοικονομική υποστήριξη για την ταχεία εφαρμογή διαρθρωτικών ε, μεταρρυθμίσεων και της ενίσχυσης της βιώσιμης ανάπτυξης. Κυρίε και κύριοι. Κυρίε και κύριοι. Εγώ δεν αποφασίζω τις διαδικασίες του Κοινοβουλίου. Κλείνοντας, αφήστε τον κύριο Επίτροπο να κλείσει την ομιλία του. Ο κανονισμός προβλέπει παρέμβαση του Επιτρόπου. Ας τον αφήσουμε να ολοκληρώσει παρακαλώ. The new system... Uh, Το νέο σύστημα ευθυγραμμίζεται πλήρως με την κοινωτική μέθοδο και θα αξιοποιήσει τις υπάρχουσες διαδικασίες εποπτείας, θα συνδυάσει την καλύτερη ολοκλήρωση των οικονομικών πολιτικών με χρηματοοικονομική υποστήριξη και ως εκ τούτου θα σεβαστεί τις αρχές για περισσότερη ευθύνη και δημοσιονομική πειθαρχία σε συνδυασμό με αλληλεγγύη όμως, περισσότερη αλληλεγγύη. Επίσης θα ενισχυθεί η δυνατότητα κάθε κρατός μέλους να απορροφήσει ε, ασύμετρα σοκ και θα μας βοηθήσει στην αρχική φάση προκειμένου να ενισχύσουμε την ε, δημοσιονομική μας ικανότητα. Επιπλέον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεσμεύθηκε να παρακολουθήσει με ταχύ και ε, δραστήριο τρόπο και να εφαρμόσει το σχέδιο δράσης για την καταπολέμηση της ε, φοροαποφυγής και φοροδιαφυγής ε, εν των σχετικών οδηγιών. Και στο σχέδιο δράσης περιλαμβάνονται κάποια μέτρα και δράσεις και για θέματα κοινωνικής πολιτικής και απασχόλησης. Θα προσταθούν κάποια στοιχεία στα πρακτικά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και κυρίως η γενική δέσμευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Προέδρου της. Και φαντάζομαι ότι με τη δήλωση αυτή εξασφαλίζεται σαφήνεια και ενάργεια για τις προθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θεωρώ ότι αποσαφηνίστηκαν οι προθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ευελπιστώ ότι θα υπερψηφίσετε το διπλό πακέτο εγκαίρως πριν τη διάσκεψη κορυφής ε, αυτής της εβδομάδας, γιατί θα είναι πολύ σημαντικό για την ανάκτηση της, ε, εμπιστοσύνης, της οικονομικής εμπιστοσύνης στην Ευρώπη. Θα είναι σημαντικό βήμα προόδου προς την υλοποίηση του κοινού μας στόχου για μια ε, γνήσια και βαθιά ΟΝΕ που θα εξυπηρετήσει όλους τους Ευρωπαίους πολίτες. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας, την υποστήριξη αλλά και την εμπιστοσύνη σας. Ευχαριστώ. Παρακαλώ. Ας συγκεντρωθούμε τώρα στην ψηφοφορία. Έκθεση Κοζές. Τροπολογία 73. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Πρόταση επιτροπής. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Και με ονομαστική κλίση το σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Ο κύριος Λάιχτφριτ για διαδικαστικό. Είναι διαδικαστικό. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα στεναρά να σας πω ότι δεν θέλω να επικρίνω καθόλου τον τρόπο με τον οποίο προεδρεύετε, αλλά ανησύχησα γιατί πραγματικά ε, είναι εκνευριστικό και θα παρακαλούσα ε, να μην πάθουν και τίποτα οι άνθρωποι, να τους προσέξετε γιατί επιβαρύνουν το νευρικό του σύστημα. Συμφωνώ. Έκθεση Φερέρα. Τροπολογία 83. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Ψηφίζουμε την πρόταση επιτροπή Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται και με ονομαστική κλίση το σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος άρχεται η ψηφοφορία. Voto chiuso. Τέλος ψηφοφορίας. Approvato. Εγκρίνεται. Έκθεση Λάμπερτς. Τροποδολογία 3. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίνεται. Έκθεση της Επιτροπής ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται και με νομαστική κλίση το σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Διαδικαστικό. Είναι διαδικαστικό όντως. Θα ήθελα να υπενθυμίσω στους συναδέλφους σήμερα ότι είμαστε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δεν είναι αρένα για πάλι στη λάσπη. Γιατί μερικοί γελάνε, χειροκροτάν, κραυγάζουν. Παρακαλώ, λίγο σεβασμό. Εδώ είναι παλέστρα της δημοκρατίας στην Ευρώπη. Relazione... Ωραία. Έκθεση ο Κονή. Τροπολογία 3. Ποιο είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Πρόταση επιτροπή. Επιτροπής. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Και με ονομαστική κλίση σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Έκθεση Μογάν Σαχτιέ. Παρακαλώ. Κυρία Πρόεδρε, θα είμαι σύντομα, σας το υπόσχομαι. Μία διευκρίνηση θα ήθελα. Μπορεί να είναι συντακτικό το λάθος ή τυπογραφικό, γιατί στο αιτιολογική σκέψη ΣΕΗ, στη ΓΑΜΑ, λέει ότι η κρίση της ε, πίστης ε, που υπάρχει και που δημιουργεί την κρίση είναι μια ανθρωπογενής καταστροφή. Νομίζω ότι θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και να είμαστε και αξιόπιστοι απέναντι στον κόσμο. Το να λέμε ότι η διεθνής χρηματοπιστωτική κρίση είναι ε, ανθρώπινο λάθος ε, είναι πραγματικά γελίο και δείχνει και έλλειψη σεβασμού προς ε, σημαντικές γυναίκες όπως η Λάρη Κλίντον, η κυρία Ρουσέφ, ε, Άγγελα Μέρκελ, ε, Κάθριν Άστον, αν μιλούμε ότι είναι λάθος του άντρα αυτό το λάθος. Μήπως πρόκειται για την προγραφικό λάθος ή είναι απλώς γελία η διατύπωση της αιτιολογικής σκέψης γάμα. Παρακαλώ, παράγραφος 1 σε δύο τμήματα. Ποιος είναι υπέρ του πρώτου τμήματος. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 12. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Παράγραφος 13. Παράγραφος 13. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 21. Πρώτο τμήμα, ποιο είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, Ποιο είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Παράγραφος 33. Πρώτο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα, Ποιο είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Παράγραφος 35. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφος 37. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφος 57. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 63. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Αιτιολογική σκέψη α, πρώτο τμήμα. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Απορρίπτεται. Αιτιολογική σκέψη Β. Πρώτο τμήμα. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Αιτιολογική σκέψη Γ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ηλεκτρονικός έλεγχος δεν είναι σίγουρο. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Αιτιολογική σκέψη Δέλτα. Ποιο είναι υπέρ. Κανεί. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Αιτιολογική σκέψη Ι. Ποιο είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Αιτιολογική σκέψη Κάπα. Υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικό έλεγχο για την αιτιολογική σκέψη Κ. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Αιτιολογική σκέψη W. Ποιο είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Αιτιολογική... Ε, Ψηφίζουμε ε, ονομαστικά το σύνολο του νομοθετικού ψηφίσματος, άρχεται ψηφοφορία, τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Έκθεση Λιωτάρ τώρα. Παρακαλώ να σηκώνετε τα χέρια σας. Παράγραφος 7. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Παράγραφος 13. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την παράγραφο 13 άρχεται ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Παράγραφος 14. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Παράγραφος 17. Πρώτο τμήμα. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται, αλλά παρακαλώ να σηκώνετε τα χέρια σας. Δεύτερο τμήμα, ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Παράγραφος 18, ποιος είναι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 19 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 20 πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται παράγραφος 27 υπέρ κατά αποχές Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 27. Άρχεται ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 27. Ποιος είναι υπέρ. συγγνώμη, λάθος. Την 27 την ψηφίσαμε. 32. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφος 40. Υπέρ. Κατά. Ε, να σηκώνετε τα χέρια σας παρακαλώ. 40. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Σαράντα ένα υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Άρχεται η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Διαδικαστικό. Είναι πολύ, πολύ ανασχέτησαν για το 32, αλλά τους αγνοήσατε. Μπορούμε να κάνουμε ηλεκτρονικό έλεγχο για την παράγραφο 32. Παρακαλώ. Πολύ ευχαρίστως. Παράγραφος 32, ηλεκτρονικός έλεγχος, άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. εγκρίνεται που είχαμε μείνει δεύτερο τμήμα της 41 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 42 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 49 υπέρ πρώτο τμήμα κατά ηλεκτρονικός έλεγχος άρχεται ψηφοφορία Τέλος. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφος 50. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται. 51 υπέρ. Κατά Απορρίπτεται. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 51. Άρχεται ψηφοφορία. Λίγη ψηφοφορία. Απορρίπτεται. 67. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Αιτιολογική σκέψη γ. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Αιτιολογική σκέψη J, πρώτο τμήμα, Ποιο είναι υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. Αιτιολογική σκέψη K, Ποιο είναι υπέρ. Κατά, αποχές, μάλλον απορρίπτεται, αλλά αν θέλετε να το ελέγξουμε και ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Απορρίπτεται. Αιτιολογική σκέψη νη. Πρώτο τμήμα. Πέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Αιτιολογική σκέψη ο. Όμικρον. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Πι. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται μάλλον, αλλά στο ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Αιτιολογική σκέψη W. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Προτείνω, ε, ψηφίζουμε το σύνολο της πρότασης. Υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίνεται. Έκθεση Σιλβία Κώστα. Παράγραφο 20. Παράγραφος 20. Θέλετε ηλεκτρονικό έλεγχο. Καμία αντίρρηση. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την τελική ψηφοφορία της έκθεσης Λιωτάρα. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται. Έκθεση Κώστα τώρα. Παρακαλώ να σηκώνετε τα χέρια. Παράγραφος 20. Πρώτο τμήμα. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 22. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Με ονομαστική κλίση το δεύτερο τμήμα, Ποιο είναι υπέρ, ε, συγγνώμη, άρχεται η ψηφοφορία, τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται και τρίτο τμήμα με ονομαστική κλίση, άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται. 25. Πρώτο τμήμα. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Παράγραφος 30. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Παράγραφος 32. Πρώτο τμήμα, ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Παράγραφος 74. Ποιος είναι υπέρ. Κατά, αποχές, απορρίπτεται. Αιτιολογική σκέψη λάμδα. Ποιο είναι υπέρ για το πρώτο τμήμα. Κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές Απορρίπτεται το σύνολο της πρότασης τώρα. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Έκθεση Τυρολιά. Με ονομαστική κλίση ψηφίζουμε την παράγραφο 15. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Παράγραφος 17. Πρώτο τμήμα. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, ε, συγγνώμη, ονομαστική κλίση, άρχιτη ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 23. Πρώτο τμήμα. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος για το δεύτερο τμήμα. Άκτη ψηφοφορία. Τέλος. εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα. Ποιο είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Με ονομαστική κλίση τώρα το σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται και περνάμε στην έκθεση Ρώση. Παράγραφος 25. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. και το σύνολο του νομοθετικού ψηφίσματος. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Technical problem. Just a moment. Τεχνική εμπλοκή. Μια στιγμή. Try again. Doesn't work. Πάλι να δοκιμάσουμε, δεν δουλεύει το σύστημα όμως. Yes, thank you, President. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ήθελα προηγουμένως να κάνω μια διαδικαστική παρέμβαση. Χαίρομαι που ο κύριος Επίτροπος είναι ακόμα εδώ και είναι διαδικαστικό αυτό το θέμα, ενδεχομένω να ενδιαφέρει και τον κύριο Ρέν. Δεν έχω κανένα πρόβλημα με το γεγονός ότι η Κομισιόν πριν από τις ψηφοφορίες μπορεί να θέλει να κάνει μια σύντομη παρέμβαση. Σε αυτή την περίπτωση η Κομισιόν είχε να κάνει μια πολύ σημαντική παρέμβαση που ήταν και αναφερόμενη στο πολύπλοκο περιεχόμενο της ψηφοφορίας. Καλό θα ήταν να ακούσει η Κομισιόν σε αυτό που λέω. Νομίζω ότι όταν έχουμε να κάνουμε να κάνει η Κομισιόν τέτοιες παρεμβάσεις μακροσκελής πριν από την ψηφοφορία, θα πρέπει να αναφέρεται στη μέση διάταξη ότι θα υπάρξει χρόνος παρέμβασης ώστε να μπορούν να έρθουν και οι επίτροποι να έρθουν ενώπιον της Ολομέλειας. Θα μπορούσε να γίνει χθε το βράδυ, θα μπορούσε να είναι σήμερα το πρωί, να εξηγήσουν τι θέλουν. Και ελπίζω λοιπόν ότι η Κομισιόν μπορεί να το καταγράψει. Θα ήταν χρήσιμο <clears throat> αν πρόκειται για παρέμβαση 10 λεπτών και όχι ενό λεπτού μονάχα, αυτό να γίνεται εκτό τη ψηφοφορία και έτσι η άτακτη συμπεριφορά η οποία οδήγησε σε βαθιά ματέωση στους άλλους βουλευτές δεν θα μπορούσε να επαναληφθεί. Ευχαριστώ. Κυρία Φώστερ, υπήρχε μια συμφωνία μεταξύ της Κομισιόν και του Κοινοβουλίου. Και γι' αυτό ο κύριος Επίτροπος είχε το δικαίωμα να κάνει μια παρέμβαση ακόμα και αν είχε κάπως πιο μικρός κελί χαρακτήρα. Υπάρχουν πάντα όρια χρονικά τα οποία δεν υπερβαίνουν τα 10 λεπτά για παρέμβαση κομισιών. Αυτή ήταν η συμφωνία και τη σεβάστηκε ο κύριος Ρεν τη συμφωνία μας. Απόλυτα. Η κυρία Μπερές, θέλετε να παρέμβετε. Πρόεδρε, ε, ναι, δράτω με τις ευκαιρίες ε, των όσων είπε η συνάδελφος διότι ο Επίτροπος που όντως ε, παρευρίσκεται ακόμα ενώπιόν μας μακρηγόρησε και δυστυχώς ε, αποδυναμώθηκε το μήνυμα που υποτίθεται ότι έπρεπε να δώσει το Κοινοβούλιο. Αλλά η δήλωση ήταν αναπόσπαστο τμήμα της συμφωνίας και ήταν πράγματι πάρα πολύ σημαντικό να γίνει η δήλωση αυτή δημόσια ε, κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας εδώ στο Κοινοβούλιο. Καλά, ας περάσουμε στις επεξηγήσεις ψήφου τώρα. Για την έκθεση Κορέρα, το λόγο έχει ο κύριος Φόρτ.